για να αποζημιωθούν τα θύματα αυτής της καταγγελίας. Θα ήθελα να εκφράσω την ελεγγύη μου προς τους πληγέντες πληθυσμούς και πίσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφράσει την αλληλεγγύη του. Φυσικά και εμείς ανησυχούμε και εκφράζουμε την ελεγγύη μας για αυτή την θεομηνία που έπληξε την Καλαβρία. Και φυσικά σύσσωμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αισθάνεται ελεγγύη με όσου υποφέρουν αυτή τη στιγμή στην πανέμορφη περιοχή της Ιταλίας και της Ευρώπη. Το πρώτο σημείο τη ημερήσια διάταξη προβλέπει δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται και τις εξελίξεις της Δημοκρατίας της Μολδαβία. Εκ μέρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μας παρουσιάσει το θέμα ο Επίτροπο Φίλε. Έχετε το λόγο κύριε Φίλε. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτές. Όταν εξετάζουμε τις σχέσεις μας με τη Μολδαβία, νομίζω πως θα συμφωνήσουν όλοι πως έχουμε επιτύχει μεγάλη πρόοδο σε χρόνο ρεκόρ. Εσωτερικά όμως η χώρα αντιμετωπίζει προκλήσεις. Το δημοψήφισμα της 5ης Σεπτεμβρίου υποτίθεται ότι θα έλυνε το αδιέξοδο με το να αλλάξει τους κανόνες εκλογής Προέδρου. Απέτυχε. Το εάν όμως ε, θα ήταν και δημοκρατικό το δημοψήφισμα ήταν επίσης σημαντικό ερώτημα. Και αυτό ήταν κάτι που επιβεβαίωσαν οι διεθνείς παρατηρητές. Οι εκλογές ε, της 28ης Νοεμβρίου είναι εξίσου σημαντικέ για την εδραίωση της δημοκρατίας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να στέλνουμε μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση προς όλους ενδιαφερομένους. Κατόπιν όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να συνεργαστούν για να εκλέξουν και πρόεδρο και για να εκλέξουν έναν πρόεδρο ικανό να οδηγήσει τη χώρα στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Ταυτόχρονα βεβαίως θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αδιάλειπτα τις ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της μολδαβικής ε, κυβέρνησης. Να τονίσω λοιπόν κάποιες σημαντικές πτυχές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο μακράν ο μεγαλύτερος δωρητής στην ε, Μολδαβία, αλλά το Μάρτιο κινητοποιήσαμε άλλους 40 δωρητές οι οποίοι δεσμεύτηκαν να δώσουν 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2010 στο 2013 στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα 500 εκατομμύρια δικές μας δεσμεύσεις. Τους ε, τελευταίους μήνες ανταποκριθήκαμε σε κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες κυβερνήσεως με το να στείλουμε υψηλόβαθμου συμβούλου στους υπουργούς, να υποστηρίξουμε εκδημοκρατισμό και ζητήματα κράτους δικαίου, με το να οργανώσουμε τις εκλογικές διαβουλεύσεις, να αντιμετωπίσουμε την κατεπίγουσα ανάγκη μετά τις πέρσινες πλημμύρες και βεβαίως να δούμε τα της εξαγωγής κρασιού της Μολδαβίας μαζί με την κυβέρνηση της ε, Μολδαβίας ε, συνεργαστήκαμε σε έργα μικρής κλίμακας στην υπερδνηστερία, κυρίως στον τομέα τον κοινωνικό του χρόνου. Θα αρχίσουμε να εφαρμόζουμε ένα συνολικό πρόγραμμα οικοδόμησης των θεσμών. κάτι το οποίο διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή. Ο τελευταίος κύκλος διαπραγματεύσεων θα, που έλαβε χώρα 13 και 14 Οκτωβρίου επιδεικνύει και πάλι την πρόοδο των ειρευτικών συνομιλιών που κινούνται με ικανοποιητική ταχύτητα. Η βοήθειά μας έχει τη μορφή άμεσων μεταφορών στον προϋπολογισμό της χώρας καθώς από το τελευταίο τρίμηνο του 2009 37 εκατομμύρια ευρώ έχουν εκταμιευτεί στο μειακή βοήθεια και άλλα 50 θα προσθεθούν σύντομα. Από αυτά, γύρω στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν απευθείας για να βοηθούν τα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού. Και τώρα που ο πρόεδρος Μπούζεκ υπέγραψε τις σχετικές νομοθετικές αποφάσεις, Αναμένουμε να εκταμιεύσουμε σύντομα τα 40 εκατομμύρια ευρώ της πρώτης δόσης μακροοικονομικής βοήθειας. Στο ίδιο πνεύμα θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα μας που αφορά πολιτικές επαφές και τεχνικές ανταλλαγές. Σε λίγες μέρες θα συναντήσω τον Πρωθυπουργό στο Λουξεμβούργο το Νοέμβριο θα συνεδριάσει η Υποεπιτροπή Εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Μολδαβίας για να εξετάσει συστάσεις εν ώψη των διαπραγματεύσεων για μια συνολική συμφωνία ελευθεροπορίου. Επιπλέον έχουμε έναν ξεχωριστό διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προχωράμε προς μια συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών. Συνεχίζεται ο διάλογος απελευθέρωσης της βίζας που ξεκίνησε τον Ιούνιο την ερχόμενη Δευτέρα ανάλογα με το αποτέλεσμα των διερευνητικών αποστολών του Σεπτεμβρίου που έγιναν από ανεξάρτητους ειδικού. Το Συμβούλιο Εξωτερικών αναμένεται να βγάλει συμπεράσματα που θα αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Θα ακούσουμε τώρα τους ε, αγορητές εκ μέρους των πολιτικών ε, ομάδων και πρώτα εκ μέρους του ΕΛΚ θα λάβει το λόγο η κυρία Μακοβέη για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι για την ευκαιρία που έχουμε να συζητήσουμε τις δρομολογήσεις μεταρρυθμίσεις και εξελίξεις στη δημοκρατία της Μολδαβίας και την πρόοδο που πραγματοποιεί η χώρα αυτή στο δρόμο της ε, για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα αυτή έχει τηρήσει όλες τις δεσμεύσεις μέχρι στιγμής και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Ένωση το αναγνωρίζει σημειώθηκε αισθητή πρόοδο σε πολλά θέματα. Για παράδειγμα, στην απονομή τη δικαιοσύνη. Έχει ξεκινήσει η μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου. Έχει ξεκινήσει και ο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και μάλιστα το Σεπτέμβριο το Κοινοβούλιο της Μολδαβίας κύρωσε το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις ε, έχουν ε, πολύ αίσια αποτελέσματα. Έχουμε όμως εχέγγυο ότι η πρόοδος αυτή θα συνεχιστεί στο μέλλον. Μέχρι στιγμής η Μολδαβία έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο από τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει η Μολδαβία να τύχει ιδιαίτερη μεταχείρισης και να αναγνωριστούν εμπράκτος οι προσπάθειές της. Θα πρέπει να ανταμείψουμε, να ανταμείψουμε τη Μολδαβία για τις προσπάθειες που έκανε, γιατί επιβραβεύσαμε τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων για την πρόοδό τους, θα πρέπει αντίστοιχα να επιβραβεύσουμε και τη Μολδαβία. Και σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση των θεωρήσεων θα πρέπει να προχωρήσουμε, γιατί και στους τέσσερις τομείς που ζητήσαμε πρόοδο η Μολδαβία τα κατάφερε. Τις 25 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να οριστικοποιήσει το σχέδιο δράσης προκειμένου να υποφεληθεί και η Μολδαβία από την κατάργηση των θεωρήσεων. Σε ό,τι αφορά την υπερδνηστερία, θα πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε μια λύση στο θέμα της υπερδνηστερίας για να σταθεροποιήσουμε την περιοχή. Και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο προκειμένου να προωθηθεί αυτή η διαδικασία της ε, ολοκλήρωσης και της ένταξης της Μολδαβίας στην Ευρώπη. Βλέπετε πώς άλλαξε το πρόσωπο της Ανατολικής Ευρώπης την τελευταία 20 ετία. Και έχουν ξεκινήσει μεταρρυθμίσεις και στη Δυτικά Βαλκάνια. Ελπίζουμε το ίδιο να συμβεί και στη Μολδαβία. Εκ μέρους των σοσιαλιστών, το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος ε, Σέβεριν. Η δημοκρατία της Μολδαβίας έχει μία και μόνο λύση μεταξύ της ε, Ευρω... Ευρω... Ε, φιλοευρωπαϊκού χαρακτήρα και της ε, υπερδυσσεριοποίησης, δηλαδή της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ευημερίας αφενός και της στροφής προς το παρελθόν της Σοβιετικής Ένωσης αφετέρου. Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα της Μολδαβίας δεν έχει σχέση με τις εξωτερικές προκλήσεις, αλλά με τον εσωτερικό διχασμό που χαρακτηρίζει τις πολιτικές ε, δυνάμεις της χώρας αυτής. Η εσωτερική πολιτική αστάθεια στέρισε από την κυβερνώντα συνασπισμό να στραφεί περισσότερο προς την Ευρώπη. Η Μολδαβία βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής και η έκβαση των πρόωρων εκλογών θα πρέπει να οδηγήσει τη χώρα σε ένα μέλλον ευρωπαϊκού εξυγχρονισμού. Γι' αυτό καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις της Μολδαβίας να προτείνουν ένα μέλλον ευρωπαϊκού εξυγχρονισμού στην ε, χώρα και να αποφύγουν οποιαδήποτε αντιπαλότητα και αντιπαράθεση ε, επικεντρωμένη ταυτόχρονα στο όραμα της χώρας ε, να υλοποιήσει τους ευρωπαϊκούς τις στόχους και την ανταξιακή της προοπτική. Ευχαριστώ. Κύριε Σεβερίν, από τους φιλελεύθερους για δύο λεπτά ο κύριος Βάτσον. θα σας ακούσουμε κύριε Βάτσον. Πριν από 18 μήνες ε, εκπλαγήκαμε από την ε, ομότητα των γεγονότων στο Κισινάου. Μετά από λίγες εβδομάδες ε, στο βήμα μας ήρθαν οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων από τη χώρα αυτή και συμμετείχαν στις εργασίες της Ολομέλειας. Συμμεριζόμαστε τον ενθουσιασμό του λαού της ε, Μολδαβίας για ένα νέο μέλλον και με μεγάλη χαρά μάθαμε την πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα αυτή. Παρ' όλα αυτά πρέπει να συμβούν ακόμα πολλά πράγματα. Ε, θα πρέπει να διωχθούν οι δράσεις αυτών των ε, βιωτήτων. Αν ε, στις εκλογές του επόμενου βήμα, ε, μήνα επιβεβαιωθούν οι σημερινοί ηθήνοντες, υπάρχει περίπτωση η χώρα αυτή να μπορέσει να ολοκληρώσει την, το μετασχηματισμό τους. Η ελπίδα λένε ορισμένοι είναι καλό πρόγευμα αλλά ε, μη αρκετό γεύμα. Σίγουρα η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να ακολουθήσει μετά τις ε, νομικές ε, πράξεις που είναι απαραίτητες και προηγούνται αυτών των μεταρρυθμίσεων. Ε, σας συγχαίρω κύριε Φούλε και εσάς και τις υπηρεσίες σας για την προσπάθειά σας να βοηθήσετε τη Μολδαβία. Καλώς ορίζουμε το σχηματισμό της ομάδας αυτής των φίλων της Μολδαβίας και τη συνάντηση που έγινε για να βοηθηθεί η Μολδαβία να προχωρήσει. Γίνεται κάθε προσπάθεια από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσουμε αυτή την πανφτωχή χώρα να προχωρήσει ε, και να υλοποιήσει τα ευρωπαϊκά ε, δεδομένα. Και όταν κοιτάξει την επόμενη εβδομάδα το Συμβούλιο το καθεστώ των θεωρήσεων, ελπίζουμε να μα βοηθήσει να βρούμε έναν τρόπο ε, για να προχωρήσουμε τις θεωρήσεις. Όπως είπε και ένας πατέρα πατέρας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η θέληση αυτή βασίζεται στο, στη θέληση του λαού των ανθρώπων για να ενταχθούν στην Ευρώπη. Και ελπίζουμε να το δείξει αυτό ο λαός ε, την επόμενη, τον επόμενο μήνα εκλογές. Η κυρία Τατιάνα Σντανόκα ε, από τους Πράσινους. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Καλωσορίζουμε την πρόοδο της ε, Δημοκρατίας της Μολδαβίας και ελπίζουμε ότι οι επερχόμενες εκλογές θα παγιοποιήσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και το σεβασμό του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μολδαβία. Το μέλλον της ε, Μολδαβίας είναι η Ευρώπη, η ένταξη στην Ευρώπη. Όλα τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο δηλώνουν ότι είναι υπέρ της ευρωπαϊκής ε, συνεργασίας και ολοκλήρωσης. Ε, η δική μου χώρα, η Λετωνία, ε, έχει μια εμπειρία από την συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξήγησα στους πολιτικούς της Μολδαβίας ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη η ένταξή της. Θα πρέπει να ενταχθούν να οι προσπάθειες, ούτω ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ε, δικαστικές, οικονομικές ε, μεταρρυθμίσεις, να καταπολεμηθεί η διαφθορά κτλ. Ε, η κοινωνία της Μολδαβίας είναι πολυγλωσσική, υπάρχουν διαφορές και λόγω της ιστορίας της. Δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν περαιτέρω χάσματα και τομές μέσα σε αυτή την κοινωνία. Ε, νομίζω ότι τα γεγονότα της 20 28 η Ιουνίου δεν νομίζω ότι βοήθησαν την κοινωνία της Μολδαβίας. Υπάρχουν πολλοί πολίτες που έχουν διπλή υπηκότητα. Θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για να μην αντιμετωπίζονται διαφορετικά αυτοί οι πολίτες, και θα πρέπει να αποκτήσουν όλοι οι πολίτες της Μολδαβίας ε, ε, καθεστώς απαλλαγμένο από τις θεωρήσεις. Εκ μέρους των ε, συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, για 1,5 λεπτό, το λόγο έχει ο φίλος Δ. Τάνοκ. Κύριε Πρόεδρε, κανείς δεν αμφισβητεί πως η Μολδαβία έχει ακόμα πολύ δρόμο για να επιτύχει το στόχο της να ενταχθεί στην Ένωση. Ένα στόχο τον οποίο στηρίζει η ομάδα μου. Παραμένει μία από τις στοχότερες χώρες στην Ευρώπη παρά το ότι είναι στον ΠΟΕ και άρα είναι ευάλωτη στο οργανωμένο έγκλημα, την σωματεμπορία και τη διαφθορά. Επίσης εμποδίζεται από την σύγκρουση με την ρωσόφωνη αποσχιστική περιοχή της υπερδνηστερίας. Από όταν όμως έφυγαν οι κομμουνιστές πριν από 15 μήνες από την εξουσία έχει σημειώσει ουσιαστική πρόοδο. Τα κόμματα της Συμμαχίας Ευρωπαϊκής Ενοποίησης που κυβερνά αυτή τη στιγμή έδειξαν μια ικανότητα για να επιταχύνουν την ενσωμάτωση της Ένωση. Η ΔΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να ασκεί πίεση στην κυβέρνηση για περαιτέρω πρόοδο Στι οικονομικές μεταρρυθμίσεις, το κράτος δικαίου και την ορθή διακυβέρνηση. Πρέπει όμως ε, να ανταμείψουμε το Κισνόβιο, κάτι το οποίο βέβαια αναφέρθηκε αλλά, ε, από πλευράς Βίζας, αλλά εγώ θέλω να αναφέρω και το ζήτημα ε, της Euronest για να συζητήσουμε εκεί πέρα τα κοινά μας συμφέροντα. Όμως παραμένει το Euronest παραλυτό ως ε, θεσμός λόγω προβλήματος με το Κοινοβούλιο της Λευκορωσίας, ε, το οποίο δεν αναγνωρίζεται ως δημοκρατικά εκλεγμένο. Ελπίζω όμως μία μέρα όλες οι χώρες στην Ανατολική εταιρική σχέση, δηλαδή Μολδαβία, Ουκρανία και μία δημοκρατική Λευκορωσία να γίνουν υποψηφίες χώρες. Και ολοκληρώνουμε το γύρο των, αγορητών εκ μέρους των ομάδων με τον κύριο Μπέλτερ για 1,5 λεπτό εκ μέρους της Ελευθερίας ε, και της Δημοκρατίας, Ευρώπης Ελευθερίας και Δημοκρατίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή δείχνει βεβαίως πως ανησυχούμε για την δημοκρατία της ε, Μολδαβίας. Και αυτό βεβαίως είναι σημαντικό γιατί στη χώρα μου εδώ και χρόνια εκδηλώνονται σημαντικές κοινωνικές πρωτοβουλίες για να προσφέρουν μια προοπτική στην ε, νεολαία της ε, Μολδαβίας σε διάφορα χωριά. Οπότε θα πρέπει να δείξουμε το ενδιαφέρον μας ε, καθώς η Μολδαβία θα πρέπει να προχωρήσει προς μια εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ανέφερε βεβαίως και ο κύριος Επίτροπος. Και θα πρέπει να δούμε ποια είναι η πιθανή κατάληξη. Να δούμε δηλαδή ποια είναι τα σημαντικότερα προϊόντα τους. Ο ίνος που έχει βεβαίως κέρια σημασία για την ε, Μολδαβία. Οπότε έχετε πραγματικά την ευκαιρία, κύριε Επίτροπε, να κάνετε κάτι για να ακουφίσετε αυτή τη χώρα και βεβαίως υπήρχε και η πρωτοβουλία της ε, καγκελαρίου Μέρκελ που απευθύνθηκε στη Μόσχα για να καταφέρει να λύσει το ζήτημα της υπερδνηστερίας και είπε πως είναι σημαντικό για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας χωρίς όμως βεβαίως να έχει ε, υπάρξει καμία κινητικότητα ακόμα στο θέμα. Εύχομαι λοιπόν να έχετε καλή επιτυχία και να έρθει ακόμη πιο κοντά στην Ευρώπη Μολδαβία, κύριε Επιτροπή. Ευχαριστούμε κύριε Μπέλντερ. Ολοκληρώθηκε ο γύρος των ομιλητών εκ μέρου των ομάδων και θα ακούσουμε τους λοιπούς ομιλητές. Πρώτα θα λάβει το λόγο ο κύριος Ουγγουρεάνου για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε καταρχήν κύριε Επίτροπε η Μολδαβία έχει αποδείξει ότι η προσήλωσή της ε, στις ε, ευρωπαϊκές προδιαγραφές και αρχές είναι γνήσια και αυθεντική. Και είναι το καλύτερο παράδειγμα από τους ανατολικούς εταίρους για την ε, αποδοχή του κοινοτικού κεκτημένου. Και μέχρι στιγμής τα διαπιστευτήρια της Μολδαβίας την καθιστούν συμβατή με τις πρόοδους των Δυτικών Βαλκανίων. Γι' αυτό η πρόοδος θα πρέπει να αναγνωριστεί και να ενθαρρυνθεί. Η επιδείνωση των δημοκρατικών θεσμών, ακόμη και στην Ουκρανία, έχει, δίνει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην πρόοδο της Μολδαβίας ε, στην Ανατολική περιοχή. Είχαμε στις 28, ε, ελπίζουμε στις 28 Νοεμβρίου οι εκλογές να επιβεβαιώσουν την ε, πορεία της Μολδαβίας προς την ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να δώσουμε θετικά μηνύματα προς τη Μολδαβία και τους Μολδαβούς. Χιλιάδες μολδαβικές οικογένειες ε, είναι διχασμένες από το φραγμό των θεωρήσεων. Ο διάλογος για τις θεωρήσεις μας δίνει τεράστιες ευκαιρίες και θα πρέπει να περάσει επιτέλους στην επιχειρησιακή φάση. Ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της 25ης Οκτωβρίου θα προσκαλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτήσει σχέδιο δράσης για την κατάργηση των θεωρήσεων. Μία φιλοευρωπαϊκή ολοκληρωμένη Μολδαβία θα έχει θετικό αντίκτυπο σε όλη την περιοχή των ανατολικών σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ μία στενής κυβέρνηση και σοβούσες διενέξεις θα εξακολουθούν να απειλούν την ευρωπαϊκή σταθερότητα. Για ένα λεπτό, το λόγο έχει η κυρία Γιώτοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Μολδαβία αντιμετωπίζει και προχώρησε πολλές αλλαγές, οι οποίες ε, συνδέονται με ένα πολυεθνικό κράτος, με την πολιτική λύση του προβλήματος της υπερνηστερίας και την ε, ένταξη της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η φιλελευθερωποίηση του καθεστώτος των ε, θεωρήσεων είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό, γιατί έχουμε δει ότι μπορεί να δώσει καλά αποτελέσματα. Η έκδοση βουλγαρικών και ρουμανικών διαβατηρίων για τους πολίτες της Μολδαβίας είναι επικίνδυνη ιστορία. Παρότι οι αρχές στο Κισινάου δηλώνουν ότι η βοήθεια που λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διανεμηθεί σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από το, την καταγωγή τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Μολδαβία που είναι μία από τις φτωχότερες χώρες. Ο κύριος Μπουσόη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. παρακολούθησα τις θετικές εξελίξεις αυτής της χώρας και τα τελευταία χρόνια ε, υπάρχει μια δέσμευση υπέρ της Ευρώπης. Θα ήθελα να υπενθυμίσω την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και της δημόσιας διοίκησης. Πρέπει παράλληλα όμως να είμαστε και ρεαλιστές και να παρατηρήσουμε και να αναγνωρίσουμε ότι η μετάβαση προς την δημοκρατία δεν θα είναι αυρόχης ποσή στη Μολδαβία. Ε, χαίρομαι που η προσπάθεια για την απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων α, προχωρεί θα ήθελα ε, να προχωρήσουμε προς μια πλήρη εξάλληψη των θεωρήσεων στο μέλλον. Ε, η Μολδαβία στις ε, εκλογές της 28 η Νοεμβρίου θα πρέπει να περάσει ένα σημαντικό τεστ, μια σημαντική δοκιμασία και ελπίζω να περάσει αυτή τη δοκιμασία η κοινωνία της. Δεδομένου των θετικών αποτελεσμάτων των της προσπάθειας της Μολδαβίας ζητάω από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσουν να στηρίζουν την δημοκρατία της Μολδαβίας για να την ενθαρρύνουν ε, προς την ε, ευρωπαϊκή της πορεία με σκοπό τελικά να ενταχθεί 100% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μπουσό. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριο Μπιέλαν. Σα ευχαριστώ. Πριν από δέκα μέρες συμμετείχα σε μια αποστολή στη Μολδαβία μαζί με την κυρία Μακοβέη και με τον κύριο Μουσόνεν. Και μάλιστα φτάσαμε στη Μολδαβία σε μια πολύ σημαντική στιγμή, λίγες εβδομάδες μετά από το αποτυχημένο δημοψήφισμα του Σεπτεμβρίου και λίγες εβδομάδες πριν τις πολύ σημαντικές βουλευτικές εκλογές που θα γίνουν στις 27 ε, Νοεμβρίου. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η στιγμή για την ε, διαδικασία της ολοκλήρωσης και της ένταξης, γιατί δύο τρίτα του πληθυσμού είναι υπέρ της ένταξης Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τον Πρωθυπουργό Φίλατ ε, στο δρόμο αυτό της ενταξιακής πορείας της Μορδαβίας, γιατί δίνει μεγάλη μάχη για να καταπολεμήσει τη μάστιγα της διαφθοράς ε, που χαρακτηρίζει τη χώρα για πολλά, για πολλά χρόνια. Φυσικά υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα με την εκρεμή διένεξη της υπερδυστερίας. Πάντως ελπίζω ότι μετά τις εκλογές ε, του Νοεμβρίου θα συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις και γι' αυτό χρειάζεται ένα σημαντικό μήνυμα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω και το Συμβούλιο Κορυφής ε, να αποφασίσει για την απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μπιέλαν. Για δύο λεπτά το λόγο έχει η κυρία Ελένα Μπασέσκο. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω όλους όσους κατέθεσαν δυνατή αυτή τη συζήτηση. Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας απέναντι στην δημοκρατία της Μολδαβίας, ιδίω τώρα ε, την παραμονή των επερχόμενων εκλογών. Η κυβέρνηση της Συμμαχίας για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση επί ένα χρόνο έχει, έχει αποδείξει με Τρομακτικέ προσπάθειες ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει θεσμικές, πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσει. και νομίζω ότι είναι ε, ηγέτες στα πλαίσια της ε, ανατολικής εταιρική σχέσης. Μην ξεχνάτε ότι αυτό ε, συμβαίνει μετά από 8 χρόνια κομμουνιστικής διακυβέρνησης, κατά οποία τα βασικά δικαιώματα, η ελεύθερη έκφραση, η ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Όλα τα βασικά δικαιώματα παραβιάστηκαν. Αυτή η μεταρρύθμιση θα πρέπει να συνεχιστεί στη δημοκρατία της ε, Μολδαβίας, ειδικά στον τομέα της ε, δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε με αποτελεσματικότητα την ε, διαφθορά. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ανθρώπινες συνθήκες κράτησης και θεμελιώδη δικαιώματα για τους ανθρώπους. Η δημοκρατία της Μολδαβίας εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο, διέρχεται μια μεγάλη και σημαντική πολιτική κρίση. Γιατί δεν επικυρώθηκε το δημοψήφισμα και δεν εξελέγει ένας πρόεδρος. Οι πρόορες εκλογές της 28ης Νοεμβρίου είναι ένα τεράστιο στίχημα για την ευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας. Η δημοκρατία θα περάσει από αυτή τη σκληρή δοκιμασία. Θα ήθελα να διατρανώσω με όλη την ευθύνη που αισθάνομαι ότι η αποτυχία της δημοκρατίας κατά τις εκλογές θα είναι μια αποτυχία της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χώρα αυτή. Χρειαζόμαστε έναν εταίρο όπου οι αξίες μας θα πριτανεύουν. Ε, γιατί είναι μια όμορη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ε, η γλώσσα που μιλάνε οι πολίτες της Μολδαβίας είναι σήμερα επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Γι' αυτό θα πρέπει ακόμα περισσότερο να τη βοηθήσουμε. Ο κύριος Βιγγενίν. <clears throat> Για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συναδελφοί. Χαίρομαι για το το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφιέρωσε χρόνο και προσοχή στην Μολδαβία, που είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Πρέπει να πω λοιπόν ε, πως ε, ο συνασπισμός που κυβερνά ο συνασπισμός για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση έκανε πάρα πολλά και ανάλογα θα πρέπει να αξιολογηθεί. Ταυτόχρονα οι πολίτες αναμένουν περισσότερα αποτελέσματα στην οικονομία και στα κοινωνικά ζητήματα. Οπότε είναι βασικό αυτό το ζήτημα. Οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάτι το στιγμίο. Πρέπει να γίνουν μια πολιτική αμετάκλητη. Το γεγονό ότι δεν αλλάζει η κατάσταση οδήγησε σε μια πολιτική αστάθεια η οποία κινδυνεύει να επαναληφθεί μετά τις εκλογές οι οποίες θα γίνουν. Οπότε η έκκλησή μου προς πολιτικές δυνάμεις ανεξαρτήτως από το αποτέλεσμα των εκλογών είναι να κάνουν ό,τι είναι αναγκαίο για να εγγυηθούν την πολιτική σταθερότητα για να εργαστούν προς το συμφέρον των πολιτών και της ευρωπαϊκής προοπτικής χώρας. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω τον κύριο Πορέμπα. Οπότε, αν στάσει αργότερα θα του δώσω το λόγο. Προς το παρόν θα δώσω το λόγο για δύο λεπτά στον κύριο Πρέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο ρουμανικός υπεριαλισμός είναι ο όρος που χρησιμοποιεί ο μολδαβικός κομμουνισμός για να μιλήσει για τη ε, στάση των Ρουμάνων πολιτικών και την κατάσταση στο Κισινάου άσχετα για το αν πρόκειται για τον πρόεδρο Μπασέσκου ή για τους Ρουμάνους Ευρωβουλευτές. Η κυβέρνηση του Κισινάου θέλει όλοι να σιωπήσουμε. Νομίζω ότι δεν είναι δικαιολογημένη μια τέτοια στάση. Δεν θα πρέπει να σιωπήσουμε. Αντίθετα, θα πρέπει να υψώσουμε στεντόρια τη φωνή μας και να καταδείξουμε την κατάσταση στη Μολδαβία. Πολλοί Ρουμάνοι, Βούλγαροι, ε, υπήκοοι διαβιούν στην Μολδαβία. Νομίζω ότι όλοι οι υπήκοοι της Μολδαβίας θα πρέπει να χαίρουν των ίδιων δικαιωμάτων. Δεν θα πρέπει να δεχόμαστε διακριτική μεταχείριση. Θα πρέπει να αυξήσουμε την πίεση κατά του Κισινάου, γιατί εδώ και ένα χρόνο και ο κυβερνών συνασπισμός δικαιολογεί τις δράσεις του με την πορεία της ένταξης της Μολδαβίας. Δεν θα πρέπει να τα, να τα δικαιολογούμε όλα στο όνομα της ε, Ευρώπης, γιατί μπορεί να λέγεται ο κυβερνό συνασπισμός, για την ε, ευρωπαϊκή ένταξη, αλλά θα άλλαζε τίποτα αν λεγόταν ε, συνασπισμός για την ε, φιλία προς τη Ρωσία, για παράδειγμα. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις μεταρρυθμίσεις στην Μολδαβία. Πήγα την περασμένη εβδομάδα στο Κισινό και την Τυρασπόλ και βλέπω ότι η, η διαδικασία της ευρωπαϊκής ένταξης είναι ουσιαστικά ο όμοιρος της, εκλογικής, της προεκλογικής εκστρατείας πολλών ε, πολιτικών δυνάμεων. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί πολλά θα εξαρτηθούν από τις εκλογές ό,τι αφορά την ε, πορεία της ε, Μολδαβίας. Οι κομμουνιστές είναι κατά της ευρωπαϊκής ένταξης και μάλιστα πριν από ένα χρόνο μας έδειξαν αυτό που ήθελαν. Οι διαμαρτυρίες του Απριλίου έδειξαν με σαφήνεια ποιε είναι οι προσδοκίε των κομμουνιστών στο Κισινάου. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τη στάση των πολιτικών κομμάτων, αλλά ελπίζω ότι και τα πολιτικά κόμματα θα αντιληφθούν τη στάση των ψηφοφόρων. Σα ευχαριστούμε κύριε Πρέντα. Για ένα λεπτό το λόγο είχε ο κύριο Μάρεκ Σίβιτς. Θα πρέπει να διαρωτηθούμε γιατί αποδίδουμε τέτοια προσοχή σε μια χώρα που βρίσκονται πολύ κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά δεν έχει πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα. Ναι. Συζητούμε λοιπόν για την Μολδαβία, γιατί είναι μια μικρή χώρα στην οποία συγκρούονται δύο κόσμοι. Ένα κόσμο που με μεγάλη δυσκολία ξεφεύγει, προσπαθεί να ξεφύγει από το παρελθόν του, τον κόσμο δηλαδή που κάποτε συμβόλιζε η Σοβιετική Ένωση, και είναι μια χώρα που εξακολουθεί να είναι διχασμένη. Ένα τμήμα της ε, συνεχίζει να βρίσκεται υποκατοχή και η ίδια η χώρα είναι έρμεο της ε, διένεξης μεταξύ εσωτερικών ε, διχασμών και συγκρούσεων. Πρόκειται για μια φτωχή μικρή χώρα που θέλει να στραφεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θέλει να εξυγχρονιστεί και να εκδημοκρατιστεί. Είναι σαν την φυσική. Γιατί στη φυσική δεν έχει σημασία η ισχύ, αλλά που βρίσκεται ο μοχλός για να σηκώσουμε μια δύναμη, ένα βάρος. Και σίγουρα είναι μικρό το ποσοστό της ε, Μολδαβίας, αλλά αν βρεθεί ο μοχλός στο σωστό σημείο, θα μπορέσουμε να φέρουμε αυτή τη χώρα στο, στην πολύ θετική εξέλιξη. Γιατί θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτούς που θέλουν να εκδημοκρατήσουν την Μολδαβία άσχετα με το κόμμα στο οποίο ανήκουν. Θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς που προσβλέπουν σε ένα καλύτερο μέλλον και θα γίνουν οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Μου επισημαίνουν ότι ο κύριος Παπαδόπουλος σήκωσε την γαλάζια κάρτα. Δεν ξέρω Μήπως θέλει απλώς ε, να μιλήσει στο Catch the Eye mm. ή να υποβάλει πρόταση προς τον κύριο Σίβιετς. Όχι, απλώς για να μιλήσει στο Catch the Eye. Θα ήθελα και πάλι να σας υπενθυμίσω, συναδελφοί, ότι η γαλάζια κάρτα, η μπλε κάρτα, δεν είναι για το Catch the Eye, αλλά σημαίνει ότι διακόπτεται τον ομιλητή για να του υποβάλλεται ερώτηση με άλλο τρόπο θα πρέπει να δηλώνετε το ενδιαφέρον σας για να μιλήσετε στο Catch the Όχι με την μπλε κάρτα. Η μπλε κάρτα έχει συγκεκριμένο σκοπό. Τελευταίος μιλητής είναι ο κύριος Κούκαν. Θα μιλήσει για δύο λεπτά και θα ολοκληρώσουμε με τον κύριο Κούκαν το γύρο της συζήτηση για τη Μολδαβία. Ο κύριος Κούκαν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι εξελίξεις στη Μολδαβία είναι πολλά υποσχόμενες. Από ό,τι φαίνεται αυτή η χώρα θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα για όλους μας υποδειγματικό μέλος της ε, σχέσης ε, ανατολικής γειτονίας και η δε φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση παρουσίασε στους Μολδαβούς ε, πολίτες μια σαφή δημοκρατική προοπτική. Παρ' όλα αυτά η εσωτερική πολιτική κατάσταση έχει στιγματιστεί αρνητικά από τα αποτελέσματα των ανεπιτυχών πολιτικών μεταρρυθμίσεων όπως ανεπιτυχές ήταν και το δημοψήφισμα. Ελπίζω οι εκλογές να είναι επιτυχείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τονίσει πιο ενεργά την πρόοδο που έχει επιτύχει η Μολδαβία. Την ερχόμενη Δευτέρα το Συμβούλιο θα υιοθετήσει αποφάσεις για την στάση της Ένωσης ε, προς τη Μολδαβία και βεβαίω θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την πρόοδο που έχει σημειωθεί και σημαντικότερο θα πρέπει να ανοίξει ο δρόμος για την κατάργηση της θεώρησης ε, από τη Μολδαβία. Αλλά βέβαια θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Όλα αυτά εξαρτώνται από τα αποτελέσματα των εκλογών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πιο θετική στη στάση της ε, εναντί της Μολδαβίας. Πρέπει να εκφράσουμε την στήριξή μας στις φιλοευρωπαϊκές εκείνες δυνάμεις που υπάρχουν στη Μολδαβία. Η Μολδαβία θα πρέπει να γίνει μέλος της ενιαίας ευρωπαϊκής οικογένειας και πρέπει να την πείσουμε πως αυτό είναι το καλύτερο μέλλον που μπορούν να περιμένουν. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο γύρος των ομιλητών. Τώρα πέραμε στην διαδικασία Catch the Eye. Έχουν εγγραφεί 7 ομιλητές. Θα λάβουν το λόγο αυτοί 7 μόνο, κανένας άλλος. Και μόνο για ένα λεπτό, αυστηρά. Θα διακόπτω τον ομιλητή αν υπερβεί αυτό το λεπτό. Η κυρία Αντρικένα πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Μολδαβία έχει κάνει πολύ πρόοδο από το σύμφωνο Μολότοφ Ρίμπεντρο που χώρισε την Ευρώπη σε σφαίρες επιρροής και έγινε μέλος της ΕΣΔ. Σήμερα είναι μια ανεξάρτητη χώρα, ταυτόχρονα είναι μια δημοκρατική χώρα που βρίσκεται κάθοδο προς την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Οπότε σήμερα θα ήθελα να ενθαρρύνω την πολιτική τάξη της χώρας, όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις και τις εθνικές, οι εθνοτικές κοινότητες να αποφύγουν τις ε, άξιες συγκρούσεις και να προετοιμάσουν το μέλλον της ε, χώρας τους για να κατευθυνθεί αυτή η χώρα προς τους ευρωπαϊκούς της στόχους. Και τέλος, η υπερδνηστερία. Η υπερδνηστερία πρέπει να το αντικείμενο πρόσοχής μας και ξέρετε πως υπήρχε και η πρωτοβουλία της κυρίας Μέρκελ και άλλων πολιτικών ηγετών για να λυθεί αυτή η παγωμένη σύγκρουση. Σας ευχαριστώ. Κύριος Πάσκου. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε Φίλε, η Μολδαβία ε, είναι το μόνο τμήμα του, των Λατινών του λατινογενούς κόσμου εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να τη φέρουμε κοντά, όλο και πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιτρέψουμε την προσχώρησή της εφόσον ολοκληρωθούν μεταρρυθμίσει. Ο κυβερνό συνασπισμό που αντιμετωπίζει, θα αντιμετωπίσει το Νοέμβριο τι εκλογέ έχει προωθήσει και επιταχύνει το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων. Θα πρέπει λοιπόν να επιβραβεύσουμε την κυβέρνηση. Γι' αυτό θα πρέπει φυσικά να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις για να μην φτάσει σε αδιέξοδο η Μολδαβία. Φυσικά πολλά θα εξαρτηθούν και από την επίλυση της ε, σύγκρουσης της υπερδυριστερίας. Γι' αυτό θα πρέπει να θαρρυθούμε από τα, τις αναγγελίες που έγιναν στο Πότσταμ στην, στην διάσκεψη κορυφής Ρωσίας-Γερμανίας και τις δηλώσεις Ντοβίλ που έδειξαν την προθυμία της Ρωσίας να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα της υπερδυστερία. Θα πρέπει να κάνουμε το τελευταίο βήμα ώστε να επιστρέψει αυτή η Λετινογενής χώρα στην σκόλπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς το χρονόμετρο φαίνεται να χάλασε, αλλά ευτυχώς διορθώθηκε το πρόβλημα. Ευχαριστούμε κύριε Πάσκου. Το λόγο κύριος Μέρσελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο παρελθόν όταν κινούσαμε τα Βαλκάνια και το πρόβλημα του Κοσφοπεδίου ή της Βοσνίας παραβλέπαμε τη Μολδαβία. Θα έπρεπε εδώ και καιρό να έχει παίξει διαμεσολαβητικό ρόλο στη σύγκρουση Μολδαβίας και γειτόνων η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τω μεταξύ βεβαίως απορρίφθηκε η διαμεσολάβησή μας το να φύγει από αυτή την ε, κατάσταση στην οποία την ε, καταδίκασε το μετασοσιαλιστικό χάος η Μολδαβία δεν θα είναι εύκολο. Βεβαίως ε, η υπερνηστερία προσπάθησε να φύγει και να αποκτήσει ανεξαρτησία της από τη Μολδαβία και βέβαια έτσι έχει καταδικαστεί σε μια τελείως αγροτική οικονομία. Φαίνεται λοιπόν πως ε, έχουμε εδώ πέρα νέα σύγκρουση την οποία θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εμποδίσουμε και ειδικά την όξυση των σχέσεων με τη Ρουμανία. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω διαδοχικές εκλογές στη Μολδαβία και τότε είχαμε επαφές με εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και της αντιπολίτευσης και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια πνοή αλλαγή και έχουν γίνει πολλές αλλαγέ. και μάλιστα πρόσφατα ο Πρωθυπουργό ε, του Συνασπισμού είπε ότι έχουν, έχει σημειωθεί πολύ σημαντική πρόοδος και νομίζω ότι πολλά οφείλονται και στις ε, ενθαρρύνσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φάνηκε μάλιστα και από την πρόσφατη αποστολή τη ε, επιτροπή Εξωτερικών στη Μολδαβία. Φυσικά ο διχασμός της Μολδαβίας εντοπίζεται κυρίως στην υπερδυνστερία και θα πρέπει να προωθήσουμε τη διαδικασία για μια ολοκληρωμένη Μολδαβία για να αρθεί αυτός ο διχασμός και να στραφεί προς το μέλλον της η Μολδαβία. Έχουμε πρόβλημα και με την μετανάστευση, εκτός από άλλα προβλήματα που υπάρχουν. Δυστυχώς απενεργοποιήθηκε το μικρόφωνο του κ. Ξύπ. Mm-hmm. Εξαντλήστε το χρόνο σας. Το λόγο θα είχε κανονικό κύριο Παρνιό, αλλά μάλλον λάθο θα είναι, γιατί ή έφυγε από την αίθουσα και δεν τον βλέπω. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Πυρίλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τι τις περασμένες εβδομάδες εγώ πήγα στο Κισινάου στη Μολδαβία και συμμετείχα σε μια συνεδρίαση που οργάνωσε ο Υπουργός Πολιτισμού για την ολοκλήρωση και ενσωμάτωση της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδίως ε, για θέματα πολιτισμού μιλήσαμε. Ε, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη θέληση για ανάπτυξη μέσα από, μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ε, δικτύων πάσης φύσεως ε, από ηλεκτρικά δίκτυα μέχρι οτιδήποτε, ε, μέχρι και οργανώσεις ε, κοινωνικο-επαγγελματικές οι πολίτες της Μολδαβίας πραγματικά επιθυμούν την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση θέλει στο εγγύς μέλλον να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνονται τα πάντα προς αυτήν την κατεύθυνση. Κόβεται το μικρόφωνο του ομιλητή. Ο κύριος Μπρόντς. Ο αριθμός ε, των ατόμων και των χωρών που αυτή τη στιγμή λαμβάνουν σε καθαρούς ε, όρους ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή τη στιγμή στο μισό και αν μπουν χώρες σαν τη Μολδαβία θα φτάσει ίσως στα 2 τρίτα κάτι το οποίο βεβαίω θα είναι στο εις βάρος ε, των χωρών που αυτή τη στιγμή είναι καθαρής φορής αλλά και των χωρών που λαμβάνουν. Και βεβαίως μίλησαν οι συνάδελφοι για την ε, μετανάστευση και βεβαίω βεβαίως δεν μιλάμε για την νόμιμη μετανάστευση αλλά ε, ουσιαστικά για την παράνομη μετανάστευση ανθρώπων οι οποίοι θα δουλεύουν με τον ε, ελάχιστο μισθό και κάτω από πολύ κακές συνθήκες. Τέλος, το 1991 διακήρυξαν εξαρτησία της από την Σοβιετική Ένωση η Μολδαβία τώρα έναντι Αργυρίων θα παραδώσει την εξαρτησία της στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία CatchDI και περνάμε στο τελευταίο τμήμα αυτής της συζήτησης δίνοντας το λόγο στον Επίτροπο Φίλε για να σχολιάσει παρατηρήσει παρατηρήσεις των συναδέλφων. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Uh. Ε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση. Είναι επίκαιρη. Και πάνω απ' όλα υπάρχει μια ενότητα ως προς το μήνυμα που στέλνουμε και υποστήριξη προς την προσπάθεια για τη Μολδαβία. Η Δημοκρατία της Μολδαβίας βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο της ιστορίας της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθάει την κυβέρνηση για να πετύχει όσα περισσότερα μπορεί από το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Ε, τη βοήθησε ιδίω τον τελευταίο χρόνο. Οι μεταρρυθμίσεις ε, απηχούν, χωρίς εξαίρεση, τον ευρύ, το ευρύ φάσμα στόχων του σχεδίου δράσης. Η επιτυχία των μεταρρυθμίσεων είναι κρίσιμη για την επιτυχία επιτυχή πορεία της δημοκρατίας της Μολδαβίας. Σε ε, περιπτώσεις και στις 30 Σεπτεμβρίου ε, όπου η ομάδα των φίλων, όπως λέγεται, επισκέφθηκε το Κισινάου, κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Γουότσον, ε, εκφράσαμε την υποστήριξή μας για μια ε, μοντέρνα και ευημερούσα Μολδαβία. με εδαφική ενότητα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ιστορία της Ευρώπης προσφέρει ένα δίδαγμα εδώ. Ε, βρίσκεται σε μια θετική πορεία η Μολδαβία και πιστεύω ότι η χώρα θα καταφέρει να πετύχει τους αναγκαίους πολιτικούς συμβιβασμούς ούτως ώστε να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις. Εμείς από πλευράς μας, στο βαθμό του δυνατού, θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των πολιτών της Μολδαβίας και να δώσουμε την απαραίτητη εξωτερική βοήθεια στις μεταρρυθμίσεις αυτές. Θα συνεχίσουμε να τους υποστηρίζουμε για να περάσουν το, τη δοκιμασία της βιωσιμότητας α, στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Και ελπίζω επίσης ότι μετά από αυτές τις εκλογές στη Μολδαβία θα υπάρχει μια πολιτική διαδικασία όπου θα ενσωμασώνει τους, άλλου, τους πάντες ε, εστιασμένοι στην Ευρώπη προς το συμφέρον των Μολδαβών πολιτών και της Ευρώπης επίσης. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Έχουν υποβληθεί έξι προτάσεις ψηφίσματος για την ολοκλήρωση της συζήτησης. Μία από το ΕΛΚ, μία από τους φιλελεύθερους, άλλη πρόταση από την ΚΟΕ, ψήφισμα από τους